τώρα σήμερα στις 12. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη, έχουμε τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Ντεγκούχτ. Έχετε το λόγο. Thank you, uh, Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάρρευση του κτίριου στην ε, Σαβάρ στην Τάκα, στο Μπαγκλαντές, 24 Απριλίου, οδήγησε σε ένα μεγάλο σοκ όλους μας. Χάθηκαν 1.127 ζωές και ήταν πάρα πολύ οι τραυματίες, κυρίως νέες γυναίκες που εργαζόντουσαν στην, ε, στην παραγωγή ενδυμάτων. μαζί με τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή, τον κύριο Άντορ, επίσης που παρακολουθούν το θέμα αυτό, θέλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ατυχημάτων. Η κλίμακα αυτού του ατυχήματος και προηγουμένων ατυχημάτων έχει οδηγήσει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας της βιομηχανίας ενδυμάτων στον Μπαγκλαντές και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό εμπλέκει και την Ευρώπη που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μπαγκλαντές. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ενώ η σημερινή συζήτηση για προφανείς λόγους εστιάζεται στο Μπαγκλαντές, ο στόχος δεν είναι να κατανομάσουμε και να επωνυδίσουμε την χώρα αυτή. Υπάρχουν αντίστοιχες συνθήκες και σε άλλες χώρες που πρέπει και εκεί να αντιμετωπιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε ταχαίως για τον Μπαγκλαντές, εξέφρασε την αλληλεγγύη της και έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Έχουμε προχωρήσει σε μια νέα ε, στρατηγική για τα θέματα των συνθηκών στην παραγωγή, στην ε, βιομηχανία ενδυμάτων στη Νότια και Νότια-Ανατολική Ασία και δεδομένου ότι είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρος στο Μπαγκλαντές, αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στον τόπο εργασίας κάναμε μια ε, έκκληση προς την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να παρέμβει το ταχύτερο δυνατό και να εξασφαλίσει ότι συμμορφούνται οι επιχειρήσεις του Μπαγκλαντές με τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και έχουμε προσφέρει και τη δική μας βοήθεια για τα θέματα αυτά. Μπορούμε ήδη να χρησιμοποιήσουμε τα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούμε εκεί για τον στόχο αυτό και θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να συνενώσει όλους τους εμπλεκόμενους για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ασφάλειας στα εργοστάσια του Μπαγκλαντές. Εμείς ε, εξετάζουμε τη δυνατότητα ενδεχομένων ενεργειών ακόμα και μέσω του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων που το Μπαγκλαντές επωφελείται από αυτό μέσα στο σύστημα όλα εκτός από τα όπλα για να έχει προτιμησιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν και μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην αλυσίδα ε, προμήθειας των ευρωπαϊκών εταιριών σε αναπτυσσόμενες χώρες και ζητούμε και από τον Μπαγκλαντές να αντιμετωπίσει την οικονομική ανισότητα και τις συνδικές εργασίες και να έχει ένα πιο υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή εκεί. Οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς εταιρείε θα πρέπει να σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα και πρότυπα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τους και να αντιμετωπίζουν με υπεύθυνο εταιρικά τρόπο και με υπεύθυνο ως προς το περιβάλλον τρόπο αυτή την παραγωγή οι 24 εταιρείες που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη, μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν ενδύματα από τον Μπαγκλαντές, έχουν υπογράψει μια κοινή συμφωνία για κώδικα πυροπροστασίας και ασφάλειας στα εργοστάσια του Μπαγκλαντές, τα οποία τους προμηθεύουν. Στην ΤΑΚΑ η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επαφές με τους αρμόδιους αξιωματούχους και τους εκπροσώπους των ενώσεων παραγωγών ενδυμάτων για να αντιμετωπίσουν τα θέματα της ασφάλειας στον τομέα αυτό. Παρόμοιες διαβουλεύσεις έχουν γίνει και με εκπροσώπους μεγάλων ευρωπαϊκών ε, εταιριών ε, ενδυμάτων και λιανικής πώλησης για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ασφάλεια στα εργοστάσια αυτά. Είναι μια περίοδος λοιπόν έντονης ε, προσπάθειες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μπαγκλαντές. Δώσαμε ένα σαφές μήνυμα ότι το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως. Μια σημαντική και σταθερή βελτίωση των συνδικών εργασία θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να απομισθούν τι ευθύνε τους και να συνεργαστούν. Τα θέματα αυτά θα τα συζητήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών μόνη τη Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρξει μια βελτίωση και χαρήκαμε για την υψηλού επίπεδου αποστολή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας των Μπαγκλαντές που οδήγησε σε τριμερείς συναντήσεις μαζί με πρόσωπους της κυβέρνησης και των εργαζομένων. Ο στόχος είναι να αποτραπούν περαιτέρω ε, τραγωδίες με μια <clears throat> ε, αξιολόγηση και έλεγχο της ασφάλειας όλων των εργοστασίων και με δράσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα το σχέδιο, αυτό είναι μια παράταση και επέκταση του σχεδίου για την πυρασφάλεια που ενεκρίθη το Μάρτιο. Επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε μεταξύ των εργαζομένων και την κατάλληλη χρησιμοποίηση των εργαζομένων και των ανέργων εκεί. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και ως ο θεματοφύλακας των διεθνώς αποδεκτών εργασιακών προτύπων. Η κοινή δήλωση τώρα αυτή του τριμερού, της τριμερούς διαλόγου πρέπει να εφαρμοστεί και να γίνει ένα σχέδιο δράσης. Και βέβαια δεν μπορούν να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά χρειάζεται συγκεκριμένη δράση και είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τον Μπαγκλαντές και τους εταίρους μας να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και πλήρως τα διεθνή πρότυπα και να συνεργαστούμε με το Διεθνές Γραφείο Εργασία για τα θέματα αυτά. Υποστηρίζουμε και τη διμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μπαγκλαντές για να υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Περιμένουμε από τι ευρωπαϊκές εταιρείε να δείξουν ε, υπεύθυνη ε, εταιρική δράση και να τηρήσουν τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ για πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η δήλωση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει επίσης να τηρηθεί. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προσπάθειες να εξασφαλίσουν το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα προμηθειών τους, όπως αναφέρονται στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους και τις εταιρείες μας για τον στόχο αυτό. Για να επιτύχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους στόχους θα συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο με τις αρχές του Μπαγκλαντές και την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασία μα μας με το διεθνέ Γραφείο εργασία. Θα εργαστούμε με όλου του εμπλεκόμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίε των κοινωνικών εταίρων στον τομέα των κλωστοϊφαντουργικών και των ενδυμάτων. Έχουμε ήδη αρχίσει να ατενίσουμε τα επόμενα βήματα που μπορούμε να αναλάβουμε για να εξασφαλίσουμε μια πιο υπεύθυνη λειτουργία τη αλυσίδα προμήθεια των Μπαγκλαντέ και αλλού. Θα ενισχύσουμε και θα εξετάσουμε την επέκταση σχεδίων τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και <clears throat> προστασία της υγείας των εργαζομένων. Και θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν προγράμματα για ελέγχου συμμόρφωσης στις βιομηχανίες του Μπαγκλαντές. Θα συνεργαστούμε με την πυροσβεστική υπηρεσία του Μπαγκλαντές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στον τομέα αυτό και να έχουμε μια καλύτερη εκπαίδευση και προστασία της υγείας των εργαζομένων στον Μπαγκλαντές. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε την κλίμακα του προβλήματος και το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μονάχα στον Παγκλατές, ούτε στον τομέα των κλωστοεφαντουργικών και των ενδυμάτων. Τονίζει η, το πρόβλημα αυτό πόσο περισσότερα χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να δώσει σάρκα και ρωστά στο ψήφισμα του του Ιανουαρίου και να συνεργαστεί με τους ομολόγους του στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και θα υπάρξει μια τροποποίηση των ρυθμίσεων και της νομοθεσίας. Εν κατακλείδη πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Είναι ο εταίρος μας, αλλά... Αλλά πρέπει να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε μαζί τους με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση των συνδικών εργασίας στον Μπαγκλαντές και θα είμαι πολύ αυστηρός εκεί. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα ξεκινήσω έρευνες. Θέλω να είμαι πολύ σαφές σε όλα αυτά. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να είναι και μια αποδοτική διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενδυμάτων, οι μεγάλοι πελάτες των βιομηχανιών του Μπαγκλαντές πρέπει να επομιστούν τη δική τους ευθύνη. Θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αλυσίδα προμήθειάς τους. Θα κάνουμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου. Ε, ελπίζουμε να γίνει αυτό τον Ιούνιο ήδη και περιμένω από αυτούς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Έχουν ήδη ε, υπογράψει μια χάρτα για τα θέματα αυτά αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι εδώ και σίγουρα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τους προμηθευτές τους. Και τέλος, <clears throat> δεν είναι μονάχα ένα θέμα εμπορίου. Το εμπόριο θα πρέπει να σέβεται μια σειρά από βασικούς κανόνες. Είναι σημαντικό το εμπόριο για τον Μπαγκλαντές. Έχει εξασφαλίσει ότι εκατομμύρια ανθρώπων και γυναικών να έχουν βρει μια θέση εργασίας. Αλλά μας ενδιαφέρει ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να προτάσετε του εμπορίου. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Το λόγο έχουν οι αγορητές των πολιτικών ομάδων. Ξεκινώντας από το ΕΛΚ, έχετε το λόγο συνάδελφε Κάσπαρη για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που είπατε, τα τελευταία σας λόγια, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλόδεκτο που το είπατε ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληθεί με, αυτά τα, με την τρομερή αυτή τραγωδία που στήχησε τη ζωή σε πάνω από χιλιά άτομα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εφαρμογής των μέτρων. Δεν πρέπει να απλώς τονίζουμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στις ε, αλυσίδες αυτές παραγωγής που χρησιμοποιούν μονάχα τις φθηνότερες συνθήκες, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται σε επίπεδο καταναλωτών. Όταν εμείς αγοράζουμε ελαφρά πικαδία προϊόντα που είναι φανερό ότι δεν μπορούν να παράγονται σε, πραγμα... σε κανονικές, σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων που εξαρτώνται από το τομέα των κλωστοϊφαντουργικών στον Μπαγκλαντές για την επιβίωσή τους και οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν σε τοπικό επίπεδο και οι οποίοι πολλές φορές παρόλες τις δυσκολίες κερδίζουν περισσότερα χρήματα από ότι ο μέσος όρος του πολίτη των Μπαγκλαντές. Αλλά θα πρέπει να δούμε και την νομική κατάσταση που ισχύει. Υπάρχει επίσης και το πρόβλημα της εγκληματικής δραστηριότητα μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Το κτίριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν σαφές και προφανές ότι δεν ήταν κατάλληλο για τέτοιες βιομηχανικές δραστηριότητες. Επομένως δεν, έχει δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές για ένα τέτοιο εργοστάσιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι τηρείται ο νόμος και σε τοπικό επίπεδο, αλλά όλα αυτά χωρίς να τα κάνουμε με μια απεικιοκρατική υπεριαλιστική νοοτροπία. Όπως είπε και ο Επίτροπος Δεχούχτ, θα πρέπει να δώσουμε και μια χείρα βοηθείας προς το Μπαγκλαντές. Έχουμε μια εμπειρία ε, αιώνων για τα θέματα της πυροπροστασίας, για την ασφάλεια των κτηρίων. Έχουμε τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα, να τα προσφέρουμε στον Μπαγκλαντές, να βοηθήσουμε να τα εφαρμόσουν όλα αυτά και φυσικά θα πρέπει συγχρόνως να σκεφτούμε περισσότερο και για την κοινή μας πολιτική εξωτερικών θεμάτων, για την κοινή μας εμπορική πολιτική, να μπορέσουμε να δώσουμε και τη δική μας εμπειρία προς τον Μπαγκλαντές, όχι ως δάσκαλοι, αλλά ως εταίροι. Και επίσης, όπως είπε και ο κύριος Δεχούχτ, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και με τις εταιρείε, όχι μόνο την αλυσίδα προμηθειών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γίνονται οι προμήθειες αυτές με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πιο βιώσιμες, βιώσιμος και αηφόρος. Να μπορέσουμε να σταματήσουμε να λειτουργούμε μονάχα με μεγάλες αλυσίδες και να βοηθήσουμε να υπάρχουν και μικρότερη παραγωγή και να έχουμε το λεγόμενο δίκαιο εμπόριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο καταναλωτή να επιλέξει τα προϊόντα τα οποία κατά την άποψή του μπορούν να παράγονται με έναν τρόπο ο οποίο είναι ισοδίκαιος και με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μια πραγματική αλληλεγγύη η οποία θα εκφραστεί από τον Ευρωπαίο καταναλωτή για του παραγωγούς από τι χώρε αυτέ. Σα ευχαριστώ για του σοσιαλίστε και δημοκράτε. Έχετε το λόγο συνάδελφε Ντεκάιζερ για 1,5 λεπτό. Merci. Μετά τη Γερμινάλη νομίζαμε ότι είχε τελειώσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά αυτό είναι όνειρο. Μετά τα διαμάντια βαμμένα σε αίμα συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες της ανήκους της εκμετάλλευσης των εργαζομένων στο Μπαγκλατές. Το δευτέρου μεγαλύτερο εξαγωγέα ενδυμάτων στον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει δύο ψηφίσματα τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο πάνω στο θέμα του 2013. Η τραγωδία όμω ήταν τέτοια αυτή τη φορά, πάνω από χίλια θύματα που η αλυσίδα των ευθυνών καταγγέλθηκε πλέον ανοιχτά. Πρόκειται για συνοχή των εργοδοτών, των μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού, αλλά και των καταναλωτών. Είναι πρόβλημα βεβαίω έλλειψη νομοθεσία, έλλειψη ε, σωστών συμφωνιών, εμπορικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα διεθνού οργανισμού εργασία κλπ. Πολλέ φορέ όμω οι μεγάλε αυτέ καταστροφέ έχουν και τα θετικά, όπω τη Μαρσινέλ στο Βέλγιο. Προωθείται έτσι η έρευνα πάνω σε θέματα ασφάλεια των ορυχείων, για παράδειγμα. Μετά το Σεβέζο, το 1976, στον τομέα τη ε, χημία. Το Σεβέζο οδήγησε στη γνωστή ομώνυμη οδηγία. Το δράμα τη Ντάκα ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε κάτι θετικό. Ξέρω ότι ήδη ελήφθησαν μέτρα σε νομοθετικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου, σε επίπεδο σχεδίων δράσης, σε επίπεδο συμφωνία όσον αφορά τι συνθήκε εργασίας με τι ξένες εταιρείε του Μπαγκλαντέ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα. Έχουμε ευθύνη και παραλαμβάνω, όπως είπα και χθε, ότι οι μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες βασίζονται στις πολιτείες δεν συνυπέγραψαν αυτήν την συμφωνία και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας στην ε, συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις ελεύθερες συναλλαγές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για την Άλντε έχετε το λόγο συνάδελφε Μπένιον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Να εκφράσω καταρχήν και εγώ την λύπη μου και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Δεν χάσαν μόνο τους οικείους τους, αλλά και τους ανθρώπους που εξασφάλιζαν τον άρτον των Πρέπει να ενισχυθούν από το κράτος δεδομένων των συνθήκων, όπως θα κάνουμε και εμείς. Άλλη μια τραγωδία λοιπόν, λίγους μήνες μετά από την φωτιά στο γνωστό εργοστάσιο. Αν τηρούνται οι αυτό μας είπαν και οι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δυστυχώ όμω δεν έγινε τίποτα. Χαίρομαι τουλάχιστον που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ αντέδρασε ταχύτερα και θέσπισε μεταρρυθμίσει, ε, σταματά ελέγχων, επιθεωρήσεων, αμοιβών. Πρέπει όμω να διασφαλίσουμε ότι αυτέ οι μεταρρυθμίσει θα υλοποιηθούν στην πράξη και ότι δεν θα παραμείνουν κενό γράμμα. Χαίρομαι επίση για τον νέο νόμο για την ασφάλεια που υπέγραψαν Ευρωπαίοι προμηθευτέ. Κρίμα όμω πολλές εταιρείες δεν συνυπέγραψαν, κυρίως αμερικανικές εταιρείε και μια μεγάλη γερμανική μάλιστα η οποία αρνήθηκε να συνυπογράψει την συμφωνία. Να μην ξεχνούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα εργοστάσια αυτά τα εργοστάσια ή μάλλον με αυτά τα εργοστάσια συνεργάζονται πολλές μεγάλες αλυσίδες της δύση και δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας. Ο Επίτροπο τουλάχιστον έκανε μια περιφεστή δήλωση, αλλά θα ήθελα να μα διευκρινίσει τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να εξασφαλίσουμε μια πιο συνεκτική στάση με του Αμερικανού εταίρους μα όσον αφορά το διεθνέ εμπόριο με τον Μπαγκλαντές. Πώ θα χρησιμοποιήσουμε τη Γενική Προτιμητική Συμφωνία ω μοχλό πίεση. και συμφωνώ με το έλκο ότι δεν είναι λύση το να αποσυρθούμε απλώ από ένα γενικό όχι και να μποϊκοτάρουμε τα προϊόντα από τον Μπαγκλατέ. Διότι το Μπαγκλατέ εξαρτάται από αυτέ τι βιομηχανίε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα λοιπόν σε ποιο βαθμό, σε ποιο μέτρο θα κάνει και τι θα κάνει η Κομισιόν. Συμπερασματικά πρέπει να δράσουμε σήμερα διότι έχουν χάσει τη ζωή του υπερβολικά πολλοί άνθρωποι και πιστεύω ότι είναι εύκολο σχετικά να προλάβουμε μελλοντικέ τραγωδίες αυτού του τύπου. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Έχετε το λόγο συνάδελφε Λαμπέρτ λεπτό. Μιλώ ως επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας με σχέσεις, ε, για με την Νοτιοανατολική Ασία και τον Μπαγκλαντές. Εκφράζω και εγώ τα συλληπιτηριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων. Πριν από λίγες μέρες, τον Μπαγκλαντές μετακίνησε ένα εκατομμύριο ανθρώπου σε περιοχέ που κινδύνευαν από τυφώνα. 13 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο λόγω πεσμένων δέντρων και έγιναν και μεγάλε ζημιέ. Το λέω αυτό γιατί μπορούν να γίνουν πολλά, όπω καταλαβαίνετε, για να μειώσουμε τον αντίκτυπο μεγάλων καταστροφών, να μειώσουμε τον κίνδυνο, όταν η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών συνεργαστούν χάρη και στη διεθνή βοήθεια. Την ίδια αποφασιστική στάση πρέπει να δείξουμε και στον τομέα τη ένδυση ή των θαλασσίων μεταφορών. Στον τομέα αυτών των ενδυμάτων εργάζονται 4 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλές γυναίκες μεταξύ αυτών, που θέλουν κάθε βράδυ να πηγαίνουν στο σπίτι του με ασφάλεια, κερδίζοντας έστω ένα χαμηλό μισθό. Η απόσταση από τι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι τεράστια. Φυσικά εδώ πρέπει να ασκήσουμε όλη την πολιτική μας ε, πίεση. Υπάρχει αντίδραση. Χαίρομαι που ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εμπλέκεται και που βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί την επιρροή της. Οι κανονισμοί για την ασφάλεια και τις φωτιές απαιτεί συνεργασία μεταξύ του ελληνικού εμπορίου, των αρχών και της κυβέρνηση και δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα λόγο να μην αναφέρουμε δημόσια και να μην κατηγορήσουμε τι εταιρείε που αρνούνται να συμπογράψουν. Όπω είπαν και οι συνάδελφοι, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, συντονισμένη προσέγγιση και όχι αποσπασματικά μέτρα εδώ και εκεί. Δεν είναι θέμα απλώ επιθεωρήσεων. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα που συζητήσαμε όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη που πρέπει να υλοποιήσουμε στην πράξη. Εμεί πάντω δεν θα υποστηρίξουμε τι τροπολογίε ή μερικέ τουλάχιστον από αυτέ. Η πρωτοβουλία βεβαίω είναι καλή. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο των συνδικάτων, συμφωνούμε όλοι με αυτό, γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πρέπει τα συνδικάτα να έχουν κάθε ελευθερία να οργανώνονται και πρέπει βεβαίω να λάβουν τι ευθύνε του και οι εργοδότε. Εννοείται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η εργοδοσία απέτυχε παταγωδό. Και βεβαίω οι επιθεωρητέ πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά του ελεύθερα όπω πρέπει, χωρί παρεμβολή από την εργοδοσία. Και αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό. Επίση, η συμφωνία GSP πρέπει να αποτελέσει κίνητρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θετικά μέτρα πριν προβούμε σε πιο σκληρές ενέργειες. Εν ώψη και των ε, συμφωνιών ελευθερού εμπορίου μεταξύ με την Ινδία, η οποία έχει και αυτή ένα πολύ σημαντικό τομέα ένδυση. Ευχαριστώ για το ECR, ο κύριος Τάνοκ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, όλοι μας θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και την αλληλεγγύη στον λαό του Μπαγκλαντές για το, την τρομερή αυτή τραγωδία στην Τάκα. Και έχουμε πάνω από 150.000 ε, Βρετανούς από τον Μπαγκλαντές που έχουν χάσει πολύ τους οικείους τους σε αυτή την καταστροφή. Όπως γνωρίζουν όλοι, αυτή η καταστροφή θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αν οι ιδιοκτήτες των κτηρίων είχαν τηρήσει και είχαν συμμορφωθεί με τα πρότυπα στην νομοθεσία του Μπαγκλαντές. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλά ψηφίσματα για τον Μπαγκλαντές τους τελευταίους μήνες και μπορεί αυτή η χώρα να νομίζει ότι την έχουμε ξεμοναχιάσει και ιδιαίτερα σε αυτήν απευθενόμαστε όταν και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Η χώρα του Μπαγκλαντέ είναι μια δημοκρατία που πρέπει να υποστηριχθεί από εμά. Υπάρχουν συστημικά προβλήματα στη βιομηχανία ενδυμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις εταιρείε και από την κυβέρνηση. Αλλά μια διαδικασία ε, τιμωρητική από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε τίποτα και ιδίω μια αναστολή του καθεστώτος ε, προτιμησιακού εμπορίου δεν θα βοηθήσει κανένα, ιδιαίτερα θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους αυτούς που εξαρτώνται από τη βιομηχανία ενδυμάτων για την επιβίωσή τους. Θα πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργήσει επικοδομητικά με τις αρχές του Μπαγκλαντές σε εταιρικό επίπεδο για να βελτιώσουν οι συνθήκες εργασίας και να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και φυσικά και η ε, πολιτές ενδυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθήσουν καλύτερα την αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας και να εξασφαλίσουν πιο υψηλά στάντα στον Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την κούε. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σπάνια οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν μια τόσο ομόφωνη άποψη σε σχέση με ένα ψήφισμα. Η καταστροφή στο Μπαγκλαντέ μας συγκλώνησε όλους μας. Αλλά ασχοληθήκαμε με τους ε, μόνο ευτυχώ έξι νεκρού στο εργοστάσιο παπουτσιών στην ε, Καμπότζη που παράγει τα παπούτσια, τα αθλητικά τη ASICS που πουλούνται μόνο για 25 ευρώ στην Ευρώπη. Αυτό το ερώτημα δεν το έχει θέσει κανένα. Εμεί ω Ευρωπαίοι έχουμε και εμείς ευθύνη για όλα αυτά τα θέματα. Με την συμπεριφορά μας ως ε, καταναλωτές, με τη δράση των επιχειρήσεών μας που ασκούν τεράστια πίεση κόστου στου παραγωγού, αλλά και γιατί αποδεχόμαστε συνθήκες παραγωγής οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη από τον καταναλωτή. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Οι περισσότεροι βουλευτέ σε αυτό το κοινοβούλιο έχουν αντιδράσει στη θέση τη δική μου πολιτική ομάδα, η οποία θέλει δεσμευτικού κανόνε για την ε, δράση των ευρωπαϊκών εταιριών σε όλο τον κόσμο. Το να υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει δεχτεί το κοινοβούλιο μα ω προπόθεση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκεί. Ελπίζω ότι κάποτε αυτό θα αντιμετωπιστεί και θα σταματήσει αυτή η απάνθρωπη συμπεριφορά. Ελπίζω ότι αρχίζετε να αλλάζετε γνώμη αγαπητοί συνάδελφοι και κάνω μια έκκληση προς την Κομισιόν να αλλάξει αυτή την αντιμετώπιση και να σταματήσει αυτή η χωρίς καμία ε, χωρίς κανένα ενδιασμό εκμετάλλευση των εργαζομένων στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο άλλους Συνάδελφε Βένσον, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βέβαια. Όπως είπαν και άλλοι μιλητέ, θέλω και εγώ να πω ότι είναι τραγικό το γεγονός. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο συγκεκριμένα, για την δήλωσή του. Εκτιμούμε βαθύτατα τις ενεργειές σας. Φυσικά είναι πολύ εύκολο σε τέτοιες περιστάσεις να λέει κανείς ότι χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία. Αυτό βεβαίως δεν αμφισβητείται. Όμως στο Μπαγκλαντές ήδη υπάρχει νομοθεσία, ήδη υπάρχουν κανόνες, απλώς δεν τηρούνται. Όπως είπε και ο κύριος Τάνοκ, έχει μεγάλη σημασία να συνεργαστούμε καταρχήν με τις αρχές. Δεν είμαστε παγκόσμιος ε, νομοθέτης, ούτε δάσκαλος. Αυτό το οποίο έχει σημασία, μετά από αυτά που είπε και ο Επίτροπος, είναι ότι τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να είναι για όλους. Περί αυτού πρόκειται. Η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο άρθρο 3 λέει ότι πρέπει να δώσουμε μάχη για τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα του ανθρώπου και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σε μέτρα κατά της ανεργίας. Όλοι χωρίς καμία διάκριση έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Όλοι όσοι εργάζονται έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή αμοιβή για τους ίδιους και την οικογένειά τους και μια ύπαρξη με ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αμοιβή η οποία θα ενισχύεται με άλλα ενδεχομένως μέσα κοινωνικής προστασίας. Όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα να ιδρύουν συνδικάτα για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να διατρανώσουμε αυτό το μήνυμα, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουμε συμπογράψει σε αυτήν την διακήρυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λάγκη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η μέση τιμή για ένα παντελόνι τζιν από το Μπαγκλαντές, η τιμή αγωγής είναι 6,5 ευρώ όταν μπαίνει αυτό στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτές οι χαμηλές τιμές μπορούν να επιτευχθούν μονάχα με τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping. Αλλά φυσικά το ίδιο παντελόνι τζιν πωλείται με 50, 60, ίσως και παραπάνω, μέχρι και 100 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν με μεγάλη σαφήνεια πού βρίσκεται η ευθύνη μέσα στην εμπορική αλυσίδα παραγωγής. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ώστε να υποχρεώσει το Μπαγκλαντές να τηρήσει τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας αλλά είναι απαραίτητο επίσης να ενισχυθούν περισσότερο και τα εργατικά συνδικάτα στο Μπαγκλαντές. Γιατί το απαραίτητο είναι να μπορούν να αγωνίζονται δίκαιες συλλογικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι στον Μπαγκλαντέ, αλλά επίσης και να αρνούνται να εργαστούν σε ανασφαλείς εγκαταστάσει και κτίρια χωρίς να υποστούν κυρώσει. Είναι λοιπόν ένα απαραίτητο στοιχείο της δράσης μας στον Μπαγκλαντέ να ενισχύσουμε τις ενώσει των εργαζομένων. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουν και οι επιχειρήσει μα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουν οι επιχειρήσεις προσπάθειες για να βελτιώσουν αυθόρμητα τις συνθήκες εργασίας των Μπαγκλαντές και να αποφύγουν επιπλέον τραγωδίες. Εμείς δεν μπορούμε να βασιστούμε μονάχα στην εθελοντική δράση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα επομιστούν και θα αναλάβουν την ευθύνη οι επιχειρήσεις και θα εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα. Όταν συναντήσετε λοιπόν τον Ιούνιο τους επιχειρηματίες, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να τους τονίσετε ότι πρέπει να τηρήσουν πλήρως τις κατευθυντήρες γραμμές του ΟΟΣΑ για την παραγωγή σε χώρες του τρίτου κόσμου και όχι μόνο στον Μπαγκλαντές αλλά και παντού. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο μεγάλη εισαγωγική αγορά για τον Μπαγκλατές. Ένα σωρό άνθρωποι όμως πλήρωσαν με τη ζωή τους τις απέσχες συνθήκες εργασίας. Τα θύματα γενικά είναι χιλιάδες. Η υπήρξη της ευθύνης τους εισαγωγής είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά τι θα κάνουμε με την αδιαφορία εναντί αυτού του δράματος στο οποίο είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι γυναίκες. Προσθέτω ότι η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθιών θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτή με τη σειρά τη στην ε, αντιμετώπιση του προβλήματο. Α μην ξεχνούμε όμω ότι αυτά τα μέτρα και οι πρωτοβουλίε δεν αρκούν. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται στην εκμετάλλευση τύπου 19ου αιώνα, ενώ ζούμε στον 21ο. Ο Επίτροπος υπογράμμισε την ευθύνη και τι πρωτοβουλίε του Διεθνού Οργανισμού Εργασία. Σύμφωνοι, τόνισε τον ρόλο του ΟΣΑ. Υπάρχει όμως και η ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μέχρι εδώ καλά. Όταν λέει ότι δεν είναι εμπορικό το πρόβλημα, εγώ θα ήθελα από όλα αυτά να τον καλέσω να διευκρινίσει την σκέψη του απαντώντα το εξή ερώτημα. Αν όλα τα μέτρα τα οποία ανέφερε δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα. Δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πρέπει με τη σειρά του να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα για να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις και τις χώρες τους να δώσουν τέλο στην σύγχρονη δουλεία που κατά τα άλλα εμείς καταγγέλουμε για δεύτερη φορά εμεί φέτο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Σας ευχαριστώ. Πριν συνεχιστή συζήτηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Μεξικού υπό την ηγεσία της ε,